Ζητήσει σχετικά με περιπτώσει παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου. Καμπότζη. Κεμ Σόκα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ από τις δημοτικές εκλογές τον Ιούνιο σημειώνεται σημαντική επιδείνωση των ε, συνθήκων ε, και κυρίως της εξέλιξης των αντιδημοκρατισμών στην Καμπότζη με την ε, σύλληψη του Κεμσούκα με επιθέσεις εις βάρος των ανεξάρτητων όσων και άλλα προβλήματα τα οποία κλιμακώθηκαν σε βία τον Ιούλιο του 2017. Η κατάσταση υπάρχει κινδύνο να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο χωρί ε, διεθνεί πιέσει και αντίσταση Χωρί να καταστεί σαφέ ότι δεν πρόκειται να επιδείξουμε καμιά άλλη ανοχή προ την κυβέρνηση τη Καμπότζη, ε, κινδυνεύουν οι αγωνιστέ των ανθρωπινών δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Πρέπει με μεγάλη προσοχή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της ε, των παραβιάσεων των δικαιωμάτων. Ε, έχουμε προσφέρει στην κυβέρνηση της Καμπότζης εμπορικά ε, προνόμια και ίσως θα έπρεπε να αναλογιστούμε και πάλι, αν συνεχιστεί αυτή η καταστολή, τη σχέση μας με την Καμπότζη. Κύριος Ντέιβιτ Μάρτιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώ τώρα τις τελευταίους μήνες τα πράγματα επιδεινώθηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ανατολική Ασία, όπως φαίνεται για το ότι έχουμε τρία καταπήγοντα για εκείνες τις χώρες σε μια ολομέλεια. Η Καμπότζη δυστυχώς δεν επετέλεσε εξαίρεση και με δεδομένο το παρελθόν, την πρώτη ιστορία της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τις βασικές αξίες ε, που να προστατεύονται σε αυτές τις χώρες αλλά τώρα βρίσκονται υπό δίωξη. Θα πρέπει να αποφυλακιστούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, θα πρέπει να ε, λειτουργήσουν τα πολιτικά κόμματα και να μπορεί ο κόσμος να έχει πολιτικές εκστρατείες και έτσι να γίνουν φυσιολογικές εκλογές ε, οι οποίες να μην ε, είναι νόθες 400 εκατομμύρια από το 2014 μέχρι το 2020 έχουμε διαδώσει. Έχουν πρωτομισιακές εμπορικές συμφωνίες γιατί είμαστε κοινότητα αξιών και αυτές αξίες θέλουμε να προαγάγουμε σε σχέση με αυτή τη χώρα και ελπίζουμε αυτές αξίες να τις σεβαστούν και εκεί. Πρόεδρος. Ένα λεπτό, Μαρία Κριστίν Βερζιάτ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτέ τι χώρε για τι οποίε εμεί ε, καταγγέλουμε τακτικά το ότι γίνονται παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό είναι σωστό για τα πράγματα όπω είπατε πάνε προ το χειρότερο. Πρώτα-πρώτα ε, έχουμε όλε αυτέ τι παραβιάσει τι οποίε καταγγέλουμε και ανησυχούμε για τα πολιτικά δικαιώματα και για την κοινωνική κατάσταση. Υπάρχει διαφθορά, υπάρχουν απαλωτριώσεις και 56% της γης έχει ασχεθεί και απαλωτριωθεί και φυλακίζουν πάρα πολύ, υπάρχουν εκτοπίσεις, ε, φτώχεια ε, και μάλλον περισσεύουν αυτά σε εκείνη την υπερχή του κόσμου. Υπάρχει μια καταστολή εις βάρος όλων που καταγγέλουν αυτά τα φαινόμενα με το θέμα της μετανάστευσης, γιατί θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί εκεί η μετακίνηση πληθυσμών είναι έντονο φαινόμενο. Ο πρώτος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βερζιά. Και τώρα ο επόμενος. Νότης Μαριάς. Ευχαριστώ πολύ, Mr. President, το πολιτικό κλίμα στην καμπότζη επιδεινώνεται οι διώξεις κατά της αντιπολίτευσης των ακτιβιστών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι στην ημερήσια διάταξη έχουμε επίσης καταδίκες αυθαίρετες. επομένως αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο και μάλιστα επιδεινώνεται όταν έχουμε δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού σε εκρεμείς δίκες και με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι γίνεται παρέμβαση στα θέματα της δικαιοσύνης πρέπει λοιπόν να σταματήσουν οι συλλήψεις πρέπει να λειτουργήσει ουσιαστικά το πολιτικό σύστημα πρέπει η κυβέρνηση να εγγυηθεί το κράτος δικαίου την ελευθερία του συνεταιρίζεστε και την ελεύθερη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. ταυτόχρονα πρέπει να σταματήσει η αρπαγή γης το 56% της γης ουσιαστικά έχει κατασχεθεί έχει δημευθεί έχει γίνει η διαδικασία αρπαγής. αρπαγή γης βεβαίως έχουμε σε πάρα πολλές χώρες και είναι απαράδεκτο. πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή ένωση να στείλει ένα μήνυμα προς την καμπότζη δεν μπορεί να συνεχίζεται η προτιμησιακή εμπορική συμφωνία με την καμπότζη να υπάρχουν αυτά τα προνόμια και όμως η καμπότζη να μην τηρεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και τώρα ο επόμενος ομιλητής, Πέτρας Αουστρεδίτσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία είπατε εκπρόσωπε και συνάδελφοι πρώτα πρώτα και εγώ να απευθύνω χαιρετισμού και καλωσόρισαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης που ήρθαν στο ημικύκλιο. Προσωπικά σας ευχαριστώ για τον αγώνα που δίνετε για πλουραλισμό και δημοκρατία στη χώρα σας επί τόσα χρόνια. Αυτά τα οποία έγιναν στη χώρα σας πρόσφατα μας έχουν προβληματίσει βαθιά. Αντί να εκμεταλλευτεί κανείς την ευκαιρία των επερχομένων εκλογών του 2018, αντί να επιλέξουν ε, το μονοπάτι της συμφιλίωσης της αξιοπρέπειας και των βασικών δικαιωμάτων αντί να καταπολεμηθεί η διαφθορά βλέπουμε καταστολή για τα ΜΜΕ, τα ανεξάρτητα την κοινωνία, την αντιπολίτευση όλα αυτά πρέπει άμεσα να λάβουν τέλος ο Κέμ Σόχα και οι άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι πρέπει να αποφυλακιστούν θα πρέπει να τους δοθεί αμνηστία έχουν προηγηθεί δεκαετίες δυστυχίας τώρα Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για συμφιλίωση και για καλύτερη ζωή για όλους στην Καμπότζη. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Στρεβίτσιος. Αποδέχεστε μια γαλάζια, μπλε κάρτα. Τον κύριο Τρεμός. Ευχαριστώ και θα ήθελα απλώς να ρωτήσω τον συνάδελφο από την Λιθουανία, τον κύριο Στρεβίτσιο, εάν συμφωνεί με το ότι θα μπορούσαμε του χρόνου να κάνουμε μια αποστολή σε εκλογές στην ε, ε, χώρα ως παρατηρητές, μια που πάντοτε ενισχύει οικονομικά την Καμπότζη. Ευχαριστώ για την ερώτηση και νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι στην καυτή επικαιρότητα. Όχι, δεν στείλαμε παρατηρητές στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές, αλλά έχουμε κοινοβουλευτικέ εκλογές το 18 και ελπίζουμε ότι οι εξεργείς δράσεις ε, αλλά και η αντιπροσωπή μας στην Πνομπέγκ θα πρέπει να πάνε εκεί για να είναι παρατηρητές εκεί στις εκλογές για να εξασφαλίσουμε όσο και το περισσότερο την ε, διαφάνεια. Ευχαριστώ. Thank you and... Uh, Ευχαριστώ. Τελευταίο συντάκτη, ο του Κέλαμ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπαντή, εκπρόσωπε. Θέλω να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Αστροβίτσιος και να στηρίξω την άποψή του για να αποσταλούν παρατηρητές στις εκλογές. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας εδώ σήμερα. Πριν από 11 μέρες, ο Κέμ Σόκα, ο γέτης της αντιπολίτευσης, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για προδοσία. Η Καμπότζη δεν έχει δημοκρατική αλλαγή. Έχει την ίδια κυβέρνηση τα τελευταία 30 χρόνια και πολλοί ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί καθώς και βουλευτές. Η δεύτερη ανησυχία μας είναι η καταποίηση των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης. Αναγκάστηκε να κλείσει σταθμός πριν από λίγες εβδομάδες και επιβλήθηκε τεράστια, τεράστιο φορολογικό πρόστιμο. Τι θα γίνει λοιπόν μέχρι τις επόμενες ε, εκλογές. Δεν πρέπει να υπάρχει ένας δημοκρατικός χώρος για την αντιπολίτευση έτσι ώστε εκλογές ε, που θα λάβουν χώρα να αντικατοπτρίζουν πραγματικά την επιθυμία της πλειοψηφία ε, του λαού της Καμπότζης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα εκ μέρους του ΕΛΚ ο κύριος Πόλτσακ. Παρακαλώ ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίζω τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης Καμπόζες που είναι εδώ παρόντες. Και επισημαίνω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατηγορείται ο Κεν Σόκα για εσχάτη προδοσία. Πρέπει λοιπόν να ε, τον βοηθήσουμε κατηγορείται για μια μυστική συνωμοσία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε τέτοιε παραβιάσεις του κράτους δικαίου. Πρέπει να υποστηρίξουμε την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση στην Καμπότζη, να πούμε ότι δεν δεχόμαστε τέτοιου είδου ε, μεθοδεύσεις και να αποστείλουμε μια αποστολή στην Καμπότζη. Ευχαριστώ πολύ. Catch the eye. Πέντε συνάδελφοι έχουν στήσει το λόγο. κύριο κύριος Πόσπισλ, πρώτος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να υποστηρίξω το ψήφισμα. Η κατάσταση στην Καμπότζη επιδεινώνεται διαρκώς. Το καθεστώς δεν ήταν ποτέ ούτε δημοκρατικό, ούτε κράτος δικαίου. Η δε σύλληψη του ηγέτη της αντιπολίτευσης αποτελεί και το αποκορύφωμα των όσων έχει πράξει μέχρι τώρα ο Πρωθυπουργό τη χώρα. Μάλιστα είχε απειλήσει να διαλύσει το κόμμα της αντιπολίτευσης εν των επόμενων εκλογών. Οπότε δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ανώθευτες οι εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα παρακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να αποστείλει παρατηρητές για τις εκλογές. Εάν τυχόν και διαλυθεί το κόμμα της αντιπολίτευση, πολύ φοβούμαι ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ε, ότι διεξάγει πραγματικά εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Καστάλτο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να χαιρετήσω και να καλέσω ε, τους ηγέτες της αντιπολίτευσης Καμπότης που βρίσκονται σήμερα εδώ να συνεχίσουν τους αγώνες τους, να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια για την ε, ανατροπή μιας, ε, ενός καθεστώτος ε, το οποίο είναι κατασταλτικό. Ε, ο Κέμ Σόγκα λοιπόν συλλαμβάνεται είναι άλλος ένας από τους ηγέτες αντιπολίτευσης που συλλαμβάνεται στη χώρα η οποία φαίνεται ότι συνεχίζει την πίεση εις βάρος αντιπολίτευσης. Εμείς επιβεβαιώνουμε την έκκλησή μας ώστε να αλλάξει το κλίμα εναντί της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να επιτραπεί η διεξαγωγή δημοκρατικών και ελεύθερων εκλογών. Καλούμε δε την ύπατη εκπρόσωπο να αξιολογήσει το ενδεχόμενο αποστολής αντιπροσωπείας για την ε, παροχή υποστήριξη προ την αντιπολίτευση τη Καμπότζη, ώστε να μπορέσει όχι μόνο να είναι υποψήφια στι εκλογέ, αλλά και να πιστέψει σε ένα πιθανό, σε ένα δυνατό μέλος της χώρας. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο. Φαρία. Ευχαριστώ πολύ. Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κούμου Σόκα παρά την βουλευτική του ασυλία συνελήφθη με αφαίρετες διαδικασίες τον κατηγορεί Πνομπένχα για προδοσία με ποινή που κινδυνεύει να έχει 15 με 20 χρόνια. Από την άλλη μεριά και το Εθνικό Δημοκρατικό Ινστιτούτο εκδιώχνεται από τη χώρα. Πρόκειται για μία απαράδεκτη τάση από ό,τι διαπιστώνουμε σε βάρος της αντιπολίτευσης και το είδαμε αυτό όμως και με τις εκλογές της δημοτικές που έγιναν πριν από λίγο. Τι θα γίνει λοιπόν με τις επόμενες ε, εκλογές. Δεν είναι δυνατόν εμείς να μην καταδικάσουμε την σύλληψη του κύριου Σόκα και να μην απαιτήσουμε την απελευθέρωση του αμέσως, καθώς επίσης και το σεβασμό του κράτους δικαίου και των δημοκρατικών ε, κανόνων. Η κυρία Σόιντροβα έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θέλω να δηλώσω περίφραστα ότι τάσομαι κατά της σύλληψης και φυλάκης του Κέμ Σόκα και βεβαίως κατά των διώξεων εις βάρος όλων των μελών του κόμματός του αλλά και κατά της καταστολής εις βάρος των, της ελευθεροτυπίας. Άκανθο στον οφθαλμό του Πρωθυπουργού είναι το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο οποίος ε, Πρωθυπουργός προσπαθεί να εγκαθιδρύσει δικτατορία στην Καμπότζη, ε, μια χώρα πλούσια, μια χώρα για την οποία εύχομαι να μπορέσει να ε, περάσει σε μια ειρηνική συμβίωση ο λαός. Και καλώς βεβαίως εδώ και τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος τελευταίος ομιλητής για τη διαδικασία αυτή. Βέντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Έχει ήδη περιγραφεί η πολύ εύθραυστη κατάσταση στην Καμπότζη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε, είναι σαφές ότι ε, ενοχλεί η άνοδος της δημοσκοπήσης αλλά και ώψη των εκλογών ε, της ε, αντιπολίτευσης. Ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τις περιοχές της υπαίθρου είναι αυτό της αρπαγής γης από μεγάλες εταιρείες εκμετάλλευσης του ζαχαρότευτλου ε, από τα χέρια των γεωργών. Πέραν αυτού όμως πρέπει να γίνονται, να γίνονται σεβαστές και αρχές του κράτους δικαίου ε, και της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπατε εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντω πολύ κακή. Η προηγούμενη εβδομάδα η δημοκρατία στην Καμποτζή ήταν επίση πάρα πολύ κακή για την ελευθερία του τύπου, όπω πολλοί είπαν, αλλά ήταν και ε, κυρίω για τον κόσμο πολύ κακή. Έχουμε στι 4 Σεπτεμβρίου την ε, σύλληψη του Κιμ Κιμσόκα και επίση το κλείσιμο ε, τη σημαντική αυτή εφημερίδα μετά από πάρα πολλέ τέτοιου είδου εξελίξει στη χώρα. Συνεχίζεται η καταστολή κατά τη ελευθερία έκφραση. Έχουν κλείσει ραδιοφωνικέ σταθμοί, έχουν γίνει συλλήψει μέλων της αντιπολίτευσης και στελεχών της κοινωνίας των πολιτών. Τώρα εδώ έχουμε επικίνδυνη κλιμάκωση, οπότε βλέπουμε να περιστέλλεται η δημοκρατία, το ΤΑΚ, ε, ΜΜΕ και όλα αυτά ενώπιση των εκλογών του 2018 συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τη δικαιοσύνη κατά ε, της αντιπολίτευσης και των μη κυβερνητικών οργανών, όλα αυτά για πολιτικούς λόγους. Και όπως γνωρίζετε και όπως μάθατε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πίεση τις αρχές τους ώστε να στη άμεσα ο Κέμ Σόκα. Αυτό έγινε ήδη φέτος. Ακούστηκε η φωνή μας. Και όταν τροποποιήθηκε δύο φορές ο νόμος για τη λειτουργία των ε, κομμάτων ε, τελικά κατέληξαν στο να διαλύσουν κάποια κόμματα. Όλα αυτά αποτελούν μια μαύρωση εκ των προτέρων των εκλογών αυτό θέτει ε, σε αμφιβολία το αποτέλεσμα των εκλογών. Επίσης ξέρετε ότι έχουμε βοηθήσει τη χώρα 10 ε, εκατομμύρια για εκλογική μεταρρύθμιση. Ε, έχουμε συνεργαστεί επίσης με τις εκλογικές αρχές για να υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση, κάποιο είδους βελτίωση εκλογικών καταλόγων κλπ. Επίσης έχουμε προσφέρει τεχνική βοήθεια για την παιδεία αλλά και έχουμε αναλάβει πρωτοβουλία παρατήρησης των εκλογών. Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων ε, ε, καταλόγων και επίσης θα γίνει και αυτή η αποστολή στην χώρα όπως έγινε και τον Ιούνιο για τις ε, δημοτικές εκλογές. Έχουμε την αντιπροσωπεία στην περιοχή όπως είπατε και θα συνεργαστούμε με την ε, ε, με τη διεθνή κοινότητα για να υπάρξουν παρατηρητές στις εκλογές. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε τις αρχές τους ώστε να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχει αξιοπιστία σε αυτές τις εκλογές. Θα πρέπει ο κόσμος να εμπιστεύει το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχουμε ε, αυτές τις αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των κομμάτων Ακριβώς σε αυτό το πνεύμα θα στείλουμε τους παρατηρητές. Ελπίζουμε να έχει αξιοπιστία η διενέργεια αυτών των εκλογών και εάν συμφωνήσει η κυβέρνηση θα κάνουμε αυτή την αποστολή των παρατηρητών τον Ιούλιο του 2018. Θα είναι πολύ σημαντικές οι πολιτικές εξελίξεις, ούτω ώστε και εμείς να δούμε πώς θα ενεργήσουμε. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό. Βοήθεια όσον αφορά την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας. Έχουμε ανεπτυσιακή συνεργασία με τη χώρα στα πλαίσια πολιετούς προγράμματος 14 με 20. Παρακολουθούμε το πώς τρέχουν τα διάφορα προγράμματα και είμαστε σε συνεχή διάλογο με την κυβέρνηση. Ανθρώπινα δικαιώματα και κράτος του δικαίου είναι πολύ βασικοί παράγοντες στην ε, νοησιακή μας πολιτική και παρακολουθούμε το αν αυτά τηρούνται. Είναι κάτι μακρόπνο η ανάπτυξη της χώρας και αξιολογούμε τις εξελίξεις λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούμε να αναστείλουμε το πρόγραμμα ανάπτυξης ανά πάσα στιγμή. Βέβαια, έτσι βοηθάμε τον κόσμο και προσπαθούμε τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Γιατί ακόμα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι σε ευάλωτη κατάσταση. Θεωρούμε ότι με την αμψιακή βοήθεια θα βελτιώσουμε την κατάσταση αυτών των ανθρώπων έχουν πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές ε, με το πρόγραμμα Everything But Arms. Όλα αυτά βοηθούν την οικονομική ανάπτυξη και παρά την τεράστια γραφική απόσταση εμείς είμαστε η βασική αγορά στην οποία εξάγει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατικές εγγύησεις. Ε, εμείς επομένως χρησιμοποιούμε κάθε διάβλο ανάπτυξης και να υπάρξει αυθεντική αλλαγή. Συνεχίζουμε την συνεργασία με τις αρχές για να δρεωθεί εκεί η δημοκρατία και να υπάρξει μια ισόρροπη δίκαιη ανάπτυξη. Θέλουμε οι αρχές της χώρας να κάνουν